Κύριε Πρόεδρε Γουαλτιέρη. Α, ωραία, όλα εντάξει, ναι. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι μια ευκαιρία για μένα να εκφράσω την ε, πολιτική μου, τα πολιτικά μου κίνητρα για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την ακρόαση αυτή. Μας ενδιαφέρει όλους να μπορέσουν όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθούν σε ισορροπία με τη φύση τους. Θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται μέσα σε μια οικονομία η οποία είναι βιώσιμη και δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι απόκληρη. Μια ανοιχτή κοινωνία, μια κοινωνία η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, αν με επικυρώσετε ως, ε, ως, ως επίτροπο, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έχω κάνει σε όλη μου την πολιτική καριέρα. Να συμβάλλω, ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να επιβληθούν στους, μικρούς. στους μικρούς. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να μην υπάρχουν άτομα τα οποία αποκλείονται από την κοινωνία είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης. Με έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι θεμητός και ισοδίκαιος μπορούν όλες οι ιδέες να ανθίσουν. Όλοι οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία της επιλογής σε ε, προσιτές τιμές. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μπορώ να έλθω ενώπιον της Επιτροπής σας. Για πρώτη φορά Ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 25 χρόνια. Ποτέ μου όμως δεν είχα φανταστεί ότι σήμερα θα βρεθώ ενώπιόν σας και φυσικά είναι μια μεγάλη τιμή για μένα και την αντιμετωπίζω με μεγάλη ταπεινοφροσύνη αυτή την τιμή. Ήμουν 21 ετών όταν μπήκα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Πολιτικού μου κόμματος στη Δανία. Το σύνθημα με το οποίο κάναμε εκστρατεία ήταν πιστεύουμε στην Ευρώπη. Και εγώ πιστεύω πράγματι στην Ευρώπη. Προχωρούμε τώρα, αν γυρίσω τρία χρόνια πίσω από σήμερα, σχεδόν ακριβώς τρία χρόνια, έγινα υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Εσωτερικών στη χώρα μου και πήγα στην πρώτη μου συνεδρίαση του Συμβουλίου Εκοφήν. Ήταν μια χρονική στιγμή μεγάλης αβεβαιότητας. Και είδα στο Συμβούλιο και ένιωσα πώς η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να γίνει μια σειρά συγκεκριμένων και πρακτικών λύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ξεπεράσαμε την θύελα της κρίσης ήταν με την αλληλεγγύη μεταξύ μας, με το να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε οι στους δε και με το να εργαστούμε για το κοινό συμφέρον. Αυτό ήταν το πνεύμα το οποίο επικράτησε στο Συμβουλιακό Κοφίν. Χάρη και στις σόφρονες αποφάσεις που πήρε η Κομισιόν, το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο, μπορέσαμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης. Ξεκινώ με αυτές τις αναμνήσεις, γιατί θέλω να μεταφέρω το ίδιο πνεύμα στην θέση, στο αξίωμα αυτό, για το οποίο είμαι υποψήφια σήμερα ενώπιόν σας. Πιστεύω ότι η προάσπιση του κοινού συμφέροντος πρέπει να είναι και ο ακρογωνίος λίθος μιας πολιτικής ανταγωνισμού. Δεν είμαι συνηθισμένη να λέω μεγάλα λόγια. Πιστεύω όμως ότι εδώ είναι πράγματι περί αυτού που πρόκειται όταν δείτε πόσο σημαντικέ είναι οι εξουσίε, οι εκτελεστικέ εξουσίε που έχει η Κομισιόν στον τομέα του ανταγωνισμού. Η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η αυστηρότητα για να εξασφαλίσουμε το κράτο δικαίου είναι απαραίτητε. Η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά την οικονομική φιλοσοφία, σε ό,τι αφορά τον νόμο. Αυτή θα είναι και η βάση για την προσωπική μου δράση. Θα είμαι ανοιχτή να ακούσω τις απόψει όλων από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τους εκπροσώπους μικρών εταιρεών. Από τα κράτη, μέλη, μέχρι τους απλούς πολίτες. Αλλά η ανάλυση του προσωπικού μου και η δική μου τελική κρίση δεν θα παρασύρεται από τις απόψεις κανενός. Το κύρος της πολιτική ανταγωνισμού και τη εφαρμογή τη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξαρτησία μα, στην αμεροληψία μα και επίση και στο σεβασμό τη εμπιστευτικότητα στην αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων. Εάν με επικυρώσετε ω Επίτροπο θα υπερασπιστώ αυτή την παράδοση αόπνος. Οι έρευνες θα γίνονται και οι αποφάσεις θα προτείνονται στο Σώμα των Επιτρόπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, από την ισχύ ή το μέγεθος μιας εταιρείας και σε περιπτώσεις κρατικής βοήθειας ανεξάρτητα από τις εμπλεκόμενες χώρες. Για μένα αυτές είναι οι κέρδιες αξίες της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού. Μεταξύ των πολλών πραγμάτων που θαυμάζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η δική σας προσήλωση σε αυτές ακριβώς τις αξίες. Εάν εγκριθώ από εσά, προσβλέπω να εργαστώ μαζί σας, να συνεργαστώ μαζί σας για να εξασφαλίσω ότι ακριβώς η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η αυστηρότητα θα είναι οι οδηγές αρχές για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Όπως σας είπα προηγουμένως, η οικονομική κρίση καταφέραμε να περιορίσουμε τις αρνητικές πτυχές της. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νιώσει την ύφεση, αυξανόμενη, την αυξανόμενη ένδια και την αβεβαιότητα για το μέλλον έχουμε ενώπιόν μας μια σαφή πρόκληση. Να επαναφέρουμε την Ευρώπη στα πόδια της. Να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης, να είμαστε καινοτόμοι, να ξαναφέρουμε μια δυναμική και κοινωνική συνοχή. Η πολιτική ανταγωνισμού έχει να διαδραματίσει ένα κέριο ρόλο στο να υποστηρίξει την έκκληση του Πρόεδρου της Κομισιόν για να υπάρξει μια ανάκαμψη σε επίπεδο απασχόλησης, μεγένθησης και επένδυση για να αντιμετωπιστούν οι συνολικέ προκλήσει για τη βιομηχανία μα, για τι μικρέ και τι μεγάλε επιχειρήσει. Ο βασικό μου στόχο λοιπόν θα ήταν να αντιμετωπίσω τα κέρια εμπόδια για την ανάπτυξη και την καινοτομία που είναι απαραίτητη για τι θέσει απασχόληση. Οι επιτυχίε των εταιριών προκύπτουν από τον θεμητό ανταγωνισμό. Σε σημαντικέ αγορέ όμω, όπω είναι η ενεργειακή και η ψηφιακή αγορά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να εξασφαλίσουμε ότι οι κυρίαρχε εταιρείε σέβονται του κανόνε του παιχνιδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και καινοτομία από μικρότερε και μεσαίε εταιρείε. Στον τομέα των κρατικών επιδοτήσεων, θα ακολουθήσω το θεματολόγιο της, του εξυγχρονισμού των κρατικών αρρωγών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν όλα τα κρατημέλη να αναλάβουν όλο και περισσότερη ενεργή ευθύνη για τις ε, κρατικές επιδοτήσεις. Θα αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η διαφάνεια και ο ανοιχτός χαρακτήρας και θα μπορέσει και το κοινό να καταλάβει πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι σπάνιοι εθνικοί πόροι. Οι πολίτες θα έχουν μια σαφέστερη εικόνα του πώς χρησιμοποιούνται τα λεφτά των φορολογουμένων. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μπορούν να είναι τμήμα μιας ευρύτερης συζήτηση ενίοτε η εφαρμογή των κρατικών αρρωγών και των κανόνων για τις συγχωνεύσεις και την ε, νομοθεσία αντιτράστ έχουν κάποιο βραχυχρόνιο, βραχυπρόθεσμο τίμημα. Ο θεμητός ανταγωνισμός και η αλλαγή στις αγορές μας έχουν εν καιρό ένα πραγματικό μέρισμα ανάπτυξης. Ένα πραγματικό μέρισμα, αλλά μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να έχουν κοινωνικό κόστος. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης για να εξασφαλίσω ότι οι παρεμβάσεις τους δεν αναχαιτίζουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Και συγχρόνως θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να εξασφαλίσω ότι τα συνοδευτικά μέτρα για αυτές τις μεταβάσεις λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνική διάσταση. Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε εδρεωμένες και υγιείς αρχές. Οι αρχές αυτές είναι σαφείς μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δοκιμαστεί από τον χρόνο. Το να κρατήσουμε την ενιαία αγορά ανοιχτή και να εξασφαλίσουμε ισότητα ανταγωνισμού, αυτή είναι η πιο άμεση στόχη της πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πετύχουμε με τον τρόπο αυτό είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό από τον ίδιο τον ανταγωνισμό. Το στόχο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Από τότε που υπήρξε η πρώτη διατύπωση των κανόνων ανταγωνισμού στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ήδη λίγο που σας λέω. Η οικονομία μας είναι τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ψηφιακή οικονομία. Αυτή η εξέλιξη και άλλες εξελίξεις μας φέρνουν ενώπιον της πρόκλησης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των αγορών για να μπορούμε να τις παρακολουθούμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ακονισμένα τα εργαλεία μας και να μπορέσουμε να προβλέπουμε τις αλλαγές στην οικονομία μας. Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο η πολιτική ανταγωνισμού παίζει ένα κέριο ρόλο για να μας βοηθήσει να έχουμε και πάλι οικονομική ανάπτυξη. Για μένα δεν είναι θέμα που αφορά μονάχα τις εταιρείε και τους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τους πολίτες, με τους ανθρώπους, με εμάς τους ίδιους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι μικρές και οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να ανταγωνιστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η πειθαρχία των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να είναι καινοτόμες και να ενισχυθούν. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού. Εγώ διαφωνώ σε αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την πολιτική ανταγωνισμού όπως χρειαζόμαστε την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις επενδύσεις, το κεφάλαιο και μια καταρτισμένη εργασιακή δύναμη. Δεν είναι μια υγιής βιομηχανική πολιτική το να προστατεύουμε εταιρείε από τον ανταγωνισμό, γιατί αυτό είναι σε βάρος των ίδιων των καταναλωτών. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού έχει μοναχικό χαρακτήρα. Κάθε άλλο. Η καλύτερη ρύθμιση δημιουργεί και υποστηρίζει την ενιαία αγορά και παροτρύνει τις εταιρείες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η ρύθμιση δημιουργεί πραγματικότητες στον τομέα της αγοράς. Το είδαμε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου είχαν μείνει εθνικές και κατακαιρματισμένες οι αγορές για πολλά χρόνια μετά την αρχική φιλελευθερωποίηση. Λένε ορισμένοι ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μια πραγματική πολιτική ανταγωνισμού όταν δεν υπάρχει πραγματική επαγρύπνηση των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαφωνώ. Ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό ανταγωνισμό είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα συνεργαστώ και με τους άλλους επιτρόπους. Είναι ένας από τους λόγους για αυτό για, που ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μοναχικό χαρτοφυλάκιο. Θέλω να συνεργαστώ και με εσά, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και άλλων επιτροπών. Θέλω όμως και σε επίσημο και σε ανεπίσημο επίπεδο να συνεργαστώ μαζί σα. Ο καθένα σα ξέρει τη δική του εκλογική περιφέρεια πολύ καλύτερα, ξέρει τι ελπίδε και τι ανησυχίε των πολιτών του καλύτερα από όλου του άλλου. Χρειάζεται να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύσει εκεί που είναι απαραίτητο να υπάρξουν ευρωπαϊκού επίπεδου λύσεις. Για να το κάνουμε αυτό, και παραθέτω αυτά που είπε ο πρόεδρο Γιούγκερ, πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και πιο φιλόδοξοι για τα μεγάλα πράγματα και πιο ταπεινοί και πιο μικροί για τα μικρά πράγματα ο συγχρονισμός <clears throat> των κρατικών επιδοτήσεων μας έχει θέσει τη σωστή τροχιά και μας βοηθάει να δούμε πού χρειάζονται οι παρεμβάσεις μας, ενώ συγχρόνως βασιζόμαστε στα κατημέλη να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν καλύτερα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τραστ, θα πρέπει να εστιάσουμε στις επιχειρηματικές πρακτικές σε κέριους τομείς. Εγώ υποστηρίζω τον στεναρό ανταγωνισμό και δεν θέλω να εμποδίσω τις μεγάλες εταιρείες από το να ανταγωνίζονται σε επίπεδο ισότητας. Δεν θα διστάσω όμως να αμφισβητήσω τη δραστηριότητα μεγάλων εταιριών όταν με καταχρηστικό τρόπο θέλουν να πιέσουν τους μικρότερους παίκτες από την αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι τις ίδιες αξίες υποστηρίζετε και εσείς. Γιατί η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι μία μορφή γραφειοκρατίας. Ακολουθεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζω, ελπίζω θα έχω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν με επικυρώσετε θα συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας και φυσικά θα είμαι προσιλωμένη σε ένα τακτικό διάλογο στα πλαίσια του ομοιβαίου σεβασμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Όχι μοναχότερα αυτό είναι επίσημα απαραίτητο, αλλά όταν είναι δυνατό. Είναι προς το συμφέρον των πολιτών και επομένως και προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εκφράζει και τους αντιπροσωπεύει. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό ξεκινάμε μια ανοιχτή, έντονη και καρποφόρα εταιρική σχέση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.